στην επόμενη συζήτηση που είναι η ανθρωπιστική κατάσταση μετά τις πρόσφατες πλημμύρες στο Πακιστάν. Εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να μας παρουσιάσει το σημείο αυτό, είναι η Κρυσταλίνα Γεωργίευα. Έχετε το λόγο για να ξεκινήσετε τη συζήτηση.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 αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειλικρινά, διότι συμπεριλάβατε το Πακιστάν στην ημερήσια διάταξη και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την ενεργή συνεισφορά του και την, την απάντηση που έδωσε, ε, διότι έχουν, ε, έχουν διοργανωθεί σε επίπεδο επίπεδο επιτροπών πολλές συνεδριάσεις και περιορίσετε το δικαίωμα ελέγχου σε μία και μόνο μέρα. Έτσι μπορέσαμε φέτος το καλοκαίρι να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για τα οικονομικά ε, πάρα πολύ γρήγορα έτσι ώστε να φύγει άμεσα η βοήθεια. Ε, ήθελα να σας ε, πω τι έχει γίνει μέχρι τώρα, να σας πω ποια είναι τα επόμενα βήματά μας, αλλά και να δούμε και ποια είναι τα μαθήματα τα οποία θα μπορούσαμε να πάρουμε και να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Καταρχά, τι έχουμε κάνει στο Πακιστάν, ποια είναι η κατάσταση στο Πακιστάν. Μία έντονη ανάμνηση που έχω είναι καταρχάς ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Έχουμε δύο καταστροφές σε μία. Στο βορρά έχουμε τρία εκατομμύρια άτομα τα οποία έχουν ε, εκτοπιστεί αν θέλετε. Ε, πρέπει να, έχουν, ε, να φύγουν, έπρεπε να φύγουν από τη χώρα τους λόγω των συγκρούσεων και τώρα τα σπίτια τους, τα καινούργια τους σπίτια καταστράφηκαν από τις πλημμύρες. Στο νότιο, στο νότο τώρα οι αγροτικές κοινότητες έχασαν όχι μόνο τα σπίτια τους αλλά και τα ζώα τους και ένα, που η κυκνοτροφία ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της ε, οικονομίας τα αριθμητικά στοιχεία όσον αφορά την καταστροφή αυτή ανεβαίνουν όλο ένα και περισσότερο. 20 εκατομμύρια Πακιστανοί έχουν πληγεί από τις πλημμύρες σε όλη τη χώρα. Πάνω από 12 εκατομμύρια άτομα ε, απαιτούν άμεση βοήθεια, υποστήριξη. Please, ε, ε, συνεχίσετε, έχετε δίκιο, ε, έχει δίκιο η Επίτροπο. θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους εκτός εθούσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει η Επίτροπος. Ξέρω ότι το θέμα το οποίο συζητούσατε προηγουμένως είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά τόσο σημαντικό είναι και το θέμα που το οποίο συζητάμε τώρα. Λοιπόν, όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία, πριν από μία εβδομάδα μιλάγαμε για 8 εκατομμύρια άτομα, τώρα ε, οι αριθμοί έχουν ε, ανέβει, είναι 12 εκατομμύρια που ζητούν άμεση βοήθεια, ε, είχαμε 8 εκατομμύρια σπίτια τα οποία είχαν καταστροφεί, τώρα ε, έχουν αυξηθεί κατά 1,5 εκατομμύρια και πάνω από 3,5 εκατομμύρια αγροτικής εκτάρια, αγροτικής γης έχουν σκεπαστεί από τα νερά. Έχουμε διάρειες, έχουμε χολέρα, ε, έχουμε επιδημίες αυτών των ασθενειών και προφανώς αυτό το οποίο χρειάζεται είναι τροφή, καθαρό νερό, ε, ε, σπίτια, τέλος πάντων θα πρέπει να προσφέρουμε κάποιο καταφύγιο στα άτομα αυτά Γι' αυτό θα ήθελα να περάσω στο επόμενο σημείο που είναι για να ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες εμείς τι κάναμε και τι πρόκειται να κάνουμε. Η ανθρωπιστική μας απάντηση ήταν σημαντική θα έλεγα. Η, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή κράτη-μέλη και κομισιό έχουν δώσει 231 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα για άμεση βοήθεια, εκ των οποίων τα 70 εκατομμύρια είναι από την Κομισιόν και τα υπόλοιπα από τα κράτη-μέλη. Τα, κράτη, τα 12 κράτη-μέλη έχουν, ε, έχουν κινητοποιήσει την ε, ενίσχυσή τους ε, μέσω του μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής θα μπορέσουμε, μπορούμε να συγκριθούμε με την έκκληση που, επίθυνε, που επίθυναν τα Ηνωμένα Έθνη και την βοήθεια που έστειλαν τα Ηνωμένα Έθνη. Βέβαια, μέσα σε μία εβδομάδα, μάλλον τα Ηνωμένα Έθνη θα απευθύνουν καινούργια έκκληση. Επίσης, στις 30 Ιουλίου ήταν σαφές ότι οι πλημμύρες θα ήταν καταστροφικές και η πρώτη μας οικονομική απόφαση, η δημοσιονομική απόφαση για 30 εκατομμύρια λήφθη στις 31 Ιουλίου, την επόμενη μέρα δηλαδή. Ενεργοποιήσαμε τον ε, μηχανισμό για αστική βοήθεια ε, στις 6 Αυγούστου με, την, ε, με, τους, με τις υπηρεσίες του Πακιστάν συγκαλέσαμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ε, που, για να συντονίσουμε τη δράση μας ε, σε συνεργασία με τις πακιστανικές αρχές έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η βοήθειά μας και ήταν η πρώτη φορά που η βοήθεια ε, των ε, κρατών μελών χρησιμοποίησε την, τις, την τις δυνατότητες αερομεταφοράς ε, που προσέφεραν οι δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, προσπαθήσαμε να στείλουμε σκηνές, φάρμακα, τροφή και υγειονομικό υλικό. Όμως παρά τις, ε, το, το, το δυναμικό και τις δυνατότητες που έχουμε αντιμετωπίζουμε ακόμα τεράστιες προκλήσεις. Καταρχάς, η ανθρωπιστική ε, κατάσταση δεν έχει λυθεί. Η κρίση υπάρχει ακόμα. Ξέρουμε από τους εθελοντές που έχουν σταλεί ότι μέχρι το Σεπτέμβριο περιμένουν 6 εκατομμύρια άτομα συμπληρωματικά, πέραν των 12 δηλαδή που ήδη χρειάζονται βοήθεια. Επομένως βλέπετε ότι η κρίση διευρύνεται όλο ένα και περισσότερο, άρα πρέπει να κινητοποιηθούμε για να μπορέσουμε να την προλάβουμε. Δηλαδή τα πράγματα θα χειροτερεύσουν πριν βελτιωθούν, κυρίως όσον αφορά τι επιδημίες. Δεύτερον, προσπαθώντας να φτάσουμε σε έναν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, ε, δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε πρώτα τα παιδιά, τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες διότι από ό,τι φαίνεται εάν δεν τους στοχεύσουμε συνειδητά κινδυνεύουν να μείνουν απ' έξω. Και αυτό προσπαθεί να κάνει η Κομισιόν συνεργαζόμενη με τους 26 εταίρους της. Τρίτον, θα πρέπει το να στέλνουμε άμεση βοήθεια. Δεν είναι θέμα απλώς και μόνο επιβίωσης, αλλά και ε, διατήρησης της σταθερότητας της χώρας ε, που αντιμετωπίζει κάποιες προκλήσεις στα θέματα ασφάλειας. Η, δυσ, δυσαρέσκεια του, κόσμου ε, εντείνεται με, την, με τα προβλήματα αυτά. Γι' αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε τα άτομα ώστε να τον περισσότερο και ώστε να τον πιο γρήγορα. Τέταρτον, είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τα άτομα βέβαια σήμερα, αλλά θα πρέπει να, ταυτόχρονα να προωθήσουμε και την ανάκαμψη. Και υπάρχουν δύο ε, προκλήσεις εδώ. Καταρχάς το θέμα, τα θέματα γεωργίας, γεωργίας. Όταν έχουμε το νερό στη διάθεσή μας θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να έχουμε το υλικό και τον εξοπλισμό επιτόπου έτσι ώστε οι γεωργοί να μπορέσουν να σπείρουν. Και δεύτερον, θα πρέπει να ε, επιδιορθώσουμε τις, ε, μετα... τις υποδομές που θα επιτρέψουν στους γεωργούς να φτάσουν στις αγορές και επίσης να ικανοποιήσουμε και τις ανάγκες των απομακρυσμένων κοινοτήτων. Μακροπρόθεσμα η χώρα αντιμετωπίζει προφανώς τεράστιες προκλήσεις όσον αφορά την ανάκαμψή της. Γίνεται μια αξιολόγηση από την Τράπεζα Ανάπτυξης και προσπαθούμε να καθορίσουμε τους μακροπρόθεσμους, τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ε, συνεργαζόμαστε με την ύπατη αρμοστή την κυρία Άστον, την κύριο Μπόμπιτη ε, ε, έτσι ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβάλει μια ολική, μια σφαιρική πρόταση για την υποστήριξη της ανάπτυξης του Πακιστάνου. τον Οκτώβριο θα υπάρξει στις 13 ε, και 14 θα υπάρχει μια συνάντηση ε, με τους εκπροσώπους του Πακιστάν και τους φίλους του Πακιστάν στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πλημμύρες στο Πακιστάν είναι ένα και μόνο στοιχείο που αποδεικνύει ότι οι κλιματικές αλλαγές θα επηρεάσουν ε, το μέλλον μας σημαντικά. Επομένως θα πρέπει να φροντίσουμε και να προλάβουμε μελλοντικές καταστροφές αλλά και να βοηθήσουμε τις χώρες να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους καταστροφές και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών. Δεν λέω ότι οι πλημμύρες αυτές είναι άμεση συνέπεια των κλιματικών αλλαγών, όμως η ένταση αυτών των καταστροφών, των φυσικών καταστροφών οφείλεται στις κλιματικές αλλαγές. Είχαμε σεισμούς στην ΑΕΤ, στην, στο Σουδάν, καταστροφές, ξηρασίες, πλημμύρες κτλ. Ε, ε, δεν έχουμε και χρήματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, ε, τα, τα ταμεία μας όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια έχουν στερέψει. Υπάρχει επίσης ένα τεράστιο χάσμα και στον, ε, στον προϋπολογισμό μας, το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όταν και εφόσον ε, πρέπει να προετοιμάσουμε και τον επόμενο ε, προϋπολογισμό. Επομένως, οι πόροι μας πρέπει να συνάδουν και με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Επίσης, από την πρώτη, μέρα της της καταστροφής είμαστε παρόντες. Όμως δεν είμαστε παρόντες στον τύπο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό θα πρέπει να βελτιώσουμε ουχή μόνο την αποτελεσματικότητά μας, αλλά και την εικόνα μας. Θα πρέπει να γίνουμε πιο ορατοί. Και αυτό φάνηκε και στη συζήτηση που είχατε και με τον πρόεδρο Μπαρόζο. Θα πρέπει να υποβάλουμε μια πρόταση στον επόμενο μήνα που θα βελτιώνει την κατάσταση. Να ολοκληρώσω αξιότιμα μέλη λέγοντας, και το λέω αυτό με ιδιαίτερη υπερηφάνεια από πλευρά των πολιτών μας, ότι το Πακιστάν μας έδειξε ότι η αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι και μόνο λόγια, αλλά είναι και πράξεις, είναι και ενέργειες και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Διότι όχι μόνο η δουλειά μας σώζει ζωές, αλλά υπερασπιζόμαστε και αξίες και αρχές που βρίσκονται στην καρδιά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ. Ε, Μιλητές εκ μέρου των πολιτικών ομάδων. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Κασμαρέκ, εκ μέρου τη ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Έχετε το λόγο κύριε συνάδελφε για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πρόκειται για βαρύτατη ανθρωπιστική καταστροφή που πλήττει δεκάδες εκατομμυρίων ανθρώπων. Θα ευχαριστήσω την Επίτροπο κυρία Γεωργίευα για την ταχεία και αποτελεσματική δράση που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κρίμα που δεν μπόρεσε να συνέλθει εκτάκτος στη διάρκεια των θερινών μηνών η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Χαίρομαι όμως που η Κομισιόν μπόρεσε και αντέδρασε και τάφθη αλληλέγγυη με τα πολλά θύματα στο Πακιστάν. Πέραν από την επίγουσα βοήθεια χρειάζεται ενίσχυση και για την γεωργία και για τις μεταφορές. Εάν δεν μπορέσει να διασωθεί η γεωργία του Πακιστάν, του χρόνου θα απειλήσει τους άμυρους αυτούς ανθρώπους νέο πλήγμα. Ίσως ωστόσο, κατά παράδοξο τρόπο, οι πλημμύρες να έχουν και ένα θετικό αποτέλεσμα, με την έννοια δηλαδή της βελτιώσεως της καταστάσεως των προσφύγων. Ελπίζω ότι θα βελτιωθούν οι ανταποκρίσεις σε τέτοιες θεομηνίες στο μέλλον και ελπίζω ότι θα βοηθήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον κυρία Ντεκάιζερ για 1,5 λεπτό επίσης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. κυρία Επίτροπε, σας συγχαίρω για την εμπλοκή σας. Ασφαλώς ανταποκριθήκατε στα καθήκοντά σας. Ωστόσο μένουν πολλά πράγματα να γίνουν. Πολλά πράγματα γιατί υπάρχει και μια απόσταση μεταξύ του Πακιστάν και της κοινή γνώμη. Οι εικόνε είναι συγκεχημένε. οι άνθρωποι δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη για να βοηθήσουν. Πρόκειται για ένα πραγματικό πρόβλημα. Ήδη βλέπετε ότι η αίθουσα του Ιμικυπρίου είναι σχεδόν κενή. Μα λένε ότι ναι, τα νερά κατεβαίνουν. Ωστόσο πρόκειται για την πιο σημαντική καταστροφή, πιο σημαντική και από το τσουνάμι. Έχω λοιπόν δύο συγκεκριμένα θέματα. Πρώτα, οι μηχανισμοί παρέμβασης. Κάνατε μεγάλες προσπάθειες και με τα κονδύλια που διαθέτατε. Δεν ε, σας κάνω καμία κριτική. Ωστόσο, η Ευρώπη έχει κάθε συμφέρον να βελτιώσει τους μηχανισμούς αυτούς ε, διάσωσης όπως βεβαίως και η Βελική Προεδρία έχει κάθε λόγο να ε, ρηχτεί στην προσπάθεια αυτή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερο, το πρόβλημα των γυναικών. Συχνά οι γυναίκες λησμονούνται ως θύματα των καταστροφών, των πολέμων. Τη στιγμή σήμερα που, μιλά, που μιλούμε υπάρχουν 300.000 γυναίκες οι οποίες πρόκειται να γεννήσουν τις επόμενες εβδομάδες 30.000 από αυτές θα χρειαστούν χειρουργικές επεμβάσεις. Κάντε σας παρακαλώ πολύ μια συγκεκριμένη ενέργεια γι' αυτό. Να βοηθήσετε τις ε, τοπικές μη κρατικέ οργανώσεις, οι οποίες είναι λίγο πολύ παρούσες παντού, η Διεθνής Οργάνωση του Planning Familia. Προσπαθήστε λοιπόν να τις βοηθήσετε και πέστε μας μετά τι έγινε δεν θα σας καταστήσουμε υπόλογοι, αλλά αναμένουμε μέσω ημών νέα από τις γυναίκες αυτές. Τώρα, εκ μέρους της ομάδας των φιλελευθέρων, ο κύριος Γκογόν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σα πω πως αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη ε, ανθρωπιστική κρίση ε, βρίσκεται, του κόσμου βρίσκεται στο Πακιστάν και το είπε η διευθύντρια της Oxfam πρόσφατα. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε λοιπόν για έναν ωκεανό προβλημάτων, δακρύων και τραγικών ιστοριών. Έχουμε καταρχήν τα, τις 20.000 ε, θύματα που δεν μπορούν 20 εκατομμύρια θύματα που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να βελτιώσουν τη θέση τους. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας έδωσε η συνθήκη της Λισαβόνας για να μπορέσουμε να παρέμβουμε αποφασιστικά. Εσείς, κύριε Επίτροπε, μας δίνετε ένα παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη όταν το επιθυμεί. Είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής και νομίζω ότι θα μπορούσαμε με τον τρόπο αυτό να εμψυχώσουμε και άλλους, να προσφέρουν κάτι στο Πακιστάν για να ξεπεράσει αυτή την αξιοθρύνητη κατάσταση. Εμείς δεν είμαστε τέλειοι βέβαια, το αναγνωρίζουμε. Νομίζω πως θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα, χωρίς να χρειαστεί να δαπανίσουμε πολύ περισσότερα. Η έκθεση Μπαρνιέ έχει ως σκοπό να πολλαπλασιαστούν τα μέσα που προσφέρουν η, η κοινότητα και τα 27 κράτη-μέλη σε περίπτωση τέτοιου είδων φυσικών καταστροφών. Τι μας προσφέρει. Καταρχήν μεγαλύτερη ορατότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι το πιο σημαντικό, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και αυτό το πλεονέκτημα. Θα πρέπει να κάνουμε την παρουσία μας πιο ορατή, γιατί είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής αυτή τη στιγμή σε ανθρωπιστική βοήθεια στον κόσμο και νομίζω θα μπορούσαμε να αναγνωριστούμε για αυτό που είμαστε, μια μεγάλη δύναμη υπέρ της ειρήνης στον κόσμο. Και το λόγο τώρα για ένα λεπτό εκ μέρους των Πρασίνων. Thank you, President. Ευχαριστώ πολύ. Όπω υπόθηκε προηγουμένω, είναι πραγματική τραγωδία τα όσα συμβαίνουν σήμερα στο Πακιστάν και χρειάζεται μακροπρόθεσμη δέσμευση που θα αναλάβουμε εμείς ενώπιον των ανθρώπων εκεί, αλλά μία δέσμευση και από την πλευρά τη ε, πρόσφατα εκλεγμένης δημοκρατικής τους ε, κυβέρνησης. για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση τέτοιου είδου καταστροφών νομίζω πως θα συμφωνήσω με την κυρία Γεώργιεβα και βεβαίως θα πρέπει να χαιρετήσουμε και την αυξανόμενη συμβολή της Ινδίας στο σχετικό ταμείο των Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω πως η διεθνής κοινότητα θα μπορούσε ε, για παράδειγμα να συγχωρέσει το διεθνές ε, χρέος του Πακιστάν για να το βοηθήσει να ξεπεράσει ε, την κατάσταση αυτή. Τρία δις ε, δόσεις δανείου κρεμούσαν την περσινή χρονιά από πλευράς Πακιστάν. Είναι δάνεια τα οποία έχει συνάψει υποδικτατορικά στρατιωτικά καθεστώτα η χώρα αυτή και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια προσπάθεια για να εξαλείψουμε τμήμα αυτού του χρέους. Νομίζω ότι καλό είναι επίσης να αναλάβουμε δράση και να πιέσουμε τους μεγάλους γεωκτήμονες του Πακιστάν να ε, συγχωρέσουν τα όσα τους χρωστούν οι ακτήμονες που τόσο σκληρά εργάζονται και που τόσο έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πλημμύρες. Madam President, Commissioner. Θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω τα σχόλια που έκανε η Επίτροπος ε, και στην Επιτροπή και εδώ, στην Ολομέλεια. Μία μάλλον η απόκριση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ημών ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστη και πρέπει να σου πω πως δράσαμε και σε διμερές επίπεδο γιατί εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο κάναμε τις προσπάθειες που μπορούσαμε. Είναι αρκετά θλιβερό το ότι Τη στιγμή που οι Πακιστανοί ζούσαν αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ο πρόεδρος τους διασκέδαζε στην Ευρώπη. Και εμείς σταθήκαμε στο πλάι τους, ε, κινητοποιηθήκαμε και είμαι ιδιαίτερα περήφανος που το κάναμε. Ε, καταστράφηκαν οι υποδομές και πρέπει να σας πω πως ο στρατός ε, ανέλαβε να τις ξαναοικοδομήσει. Ε, αυτό είναι αξιέπαινο. Όμως πριν οποιοδήποτε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σήμερα, εδώ. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν είχε προηγούμενη καταστροφή από τις πλημμύρες, χρειαζόμαστε μια χωρίς, προηγούμενη, χωρίς προηγούμενο απόκριση από πλευρά διεθνού κοινότητα. Θα πρέπει να σταθούμε δίπλα στο Πακιστάν και να βοηθήσουμε στην οικοδόμησή του να το καταλάβει αυτό ο πληθυσμό, γιατί διαφορετικά οι συνέπειε θα είναι τεράστιε. Έχουμε την αναπτυξιακή ατζέντα και εδώ θα πρέπει να τη συνδέσουμε με την εμπορική ατζέντα που θα επιτρέψουν στου πολίτε του Πακιστάν να οικοδομήσουν οι ίδιοι τη χώρα πέρα από τι προσπάθειε που θα κάνουμε εμεί. Μα ζητάνε οι πολίτε μα να γίνουμε πιο φιλόδοξοι να έχουμε ένα πλάνο ευρωπαϊκό όπως το σχέδιο Μάρσελ το οποίο ανοικοδόμησε την Ευρώπη. Αυτή είναι η διάσταση της τραγωδίας και θα σας παρακαλούσα να φανείτε αντάξει της πρόκλησης που παρουσιάστηκε. Τη παρεμβάσει εκ μέρου των πολιτικών ομάδων και ερχόμαστε στον κατάλογο των συναδέλφων που εξέφρασαν ενδιαφέρον να παρέμβουν. Ε, έχουμε τώρα ε, για 1,5 λεπτό την κυρία Στρίφλερ. Madame la Présidente, Madame Commissaire, chers... Ευχαριστώ πολύ. Η κατάσταση, η ανθρωπιστική κατάσταση στο Πακιστάν είναι δραματική. Είναι πολύ χειρότερο από το τσουνάμι το οποίο έπληξε παλαιότερα την Ασία. Και συγχαίρω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 77 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν σκοπό να βοηθήσουν του πληθυσμού που έπεσε θύμα των πλημμύρων. Και ευχαριστώ πολύ και συγχαίρω για μια φορά ακόμα την κυρία Γεώργιεβα. Πρόσβαση σε υποδομές για τα θύματα. Έχουν πλημμυρίσει τα πάντα. Έχουν καταστραφεί όλες οι υποδομές. Είναι πρωταχρικής σημασίας να δράσουμε με ουδετερότητα, με ανθρωπισμό και να βασιστούμε στις ανάγκες του πληθυσμού πριν λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση. Παρόλο που τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση τέτοιων φυσικών καταστροφών ε, έδειξαν σωστά αντανακλειστικά. Το μέγεθος της κρίσης έδειξε πως πρέπει να είμαστε πιο γρήγοροι και πιο ορατοί. Η καταστροφή αυτή υπογράμμισε μια φορά ακόμα πως είναι απαραίτητο να έχουμε τη δυνατότητα ταχείας δράσης, ταχείας επέμβασης για την πολιτική προστασία. Είναι ένα θέμα που έχω δείξει πάρα πολλές φορές, κυρία Επίτροπε. Το Νοέμβριο θα παρουσιάσετε μια ανακοίνωση για την ενίσχυση της δυνατότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκρίνεται στις φυσικές καταστροφές. Και μετά θα παρουσιάσετε και νομοθετικές προτάσεις. Εδώ λοιπόν θα παρουσιάσουμε και εμείς φιλόδοξες λύσεις. Περιμένω με ιδιαίτερη υπομονησία τις προτάσεις σας. Μαν, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή η πρόταση για τόσο πολλά εκατομμύρια βοήθειας θα πρέπει να τηρηθεί. Δεν θα πρέπει να μας τρομάξουν τα όσα μας περιμένουν. Είναι πολύ σημαντικό να συντονιστούμε μεταξύ μας στο θέμα αυτό. Και σας ρωτώ, κύριε Επίτροπε, τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Χρειάζεται περισσότερο συντονισμός μεταξύ μας. Τι πιστεύετε. Χρειάζεται ιατροφαρμακευτικό υλικό από την Ευρώπη. Πιστεύω πως ναι. Νοσηλευτές. Και αυτοί. Ανοικοδόμηση. Ναι. Πρέπει λοιπόν να βοηθηθούν οι πακιστανικές αρχές για να εξαλείψουμε τις μακροπρόθεσμες συνέπειες αυτής της καταστροφής. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τους πόρους για να στείλουμε αυτή τη βοήθεια. Ένα λεπτό επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ βεβαίως να χαιρετήσω την ε, πολύ σημαντική προσπάθεια που έχετε κάνει, κυρία Επίτροπε. Κινητοποίησαμε 230 εκατομμύρια επίγουσας βοήθειας. Είναι αξιοσημείωτο αυτό, είναι καταπληκτικό. Και η παρουσία σας εκεί αποτελεί μαρτυρία για το γεγονός πως κάνατε δικό σας το πρόβλημα θα ήθελα και εγώ να συνταχθώ με όσα είπαν οι συνάδελφοι εδώ, τα προβλήματα των γυναικών, της υγείας, όπως επίσης και τα πολιτικά προβλήματα που δημιουργούνται, γιατί βέβαια πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος ε, να περάσει ε, στο στρατόπεδο των εξτρεμιστών η χώρα αυτή. Λοιπόν, έχω πει κάτι επανειλημμένα και συγκεκριμένα μετά το σεισμό στην IT, πως πρέπει να έχουμε την δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε θέματα πολιτικής προστασίας ε, στην Ευρώπη. Η έκθεση Μπαρνιέ έχει απόλυτο δίκιο και θα ήθελα να σας πω ποιες είναι οι προθέσεις σας εκεί. Μπορείτε να μας δώσετε μια απάντηση. Ο κύριος Βαντάλεν για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στις κάτω χώρες ο αγώνας μας κατά των νερών είναι γνωστός από αιώνες. Γι' αυτό και έχουμε ιδιαίτερη συμπάθεια για τους ανθρώπους του Πακιστάν και ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας για την ανάγκη επίδειξης αλληλεγγύης και βεβαίως να μην πέσει η χώρα αυτή στα χέρια των Ταλιμπάν. Ως χριστιανός συμπάσχω και με τους Πακιστανούς χριστιανούς άκουσα από οργάνωσή τους ότι γίνονται διακρίσεις σε βάρος των χριστιανών σε ορισμένες περιοχές στην διανομή των τροφίμων. Αυτό με σοκάρισε και παρακαλώ να το λάβει υπόψη της η κυρία Επίτροπος. Ακούμε επίσης ότι οι Ταλιμπάν έχουν φωνεύσει τρεις συνεργάτες χριστιανικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο Πακιστάν. Παρακαλώ και εδώ να δείξει αλληλεγγύη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να υποστηριχθούν, πρέπει να προστατευθούν τα πρόσωπα αυτά και από τις πακιστανικές αρχές. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την συμπαράστασή μου ε, στους ανθρώπους του Πακιστάν κυρίως για την απώλεια ζώων. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Επίτροπο κυρία Γεωργίευα για την μεγάλη προσπάθεια που έχει καταβάλει για την αντιμετώπιση των δεινών του Πακιστάν. Χρειάστηκε να περάσει κάποιος χρόνος μέχρι ότου η διεθνής κοινότητα να αντιληφθεί ποιες είναι οι ανάγκες αυτές. Τώρα που το καταλαβαίνουμε καλύτερα, η ανταπόκρισή μας θα πρέπει να είναι ταχύτερη και σημαντικότερη, να προσφέρουμε περισσότερη υλική βοήθεια, ταυτόχρονα να φροντίσουμε ώστε η βοήθεια να φτάσει μέχρι όλους όσοι την χρειάζονται και οι μειονότητες. Ας μην λησμονούμε επίσης ότι το Πακιστάν βρίσκεται στην, ε, στην μεθόριο προς ε, τις ε, χώρες, προς την τρομοκρατία, ας το πω έτσι. Βέβαια, εφάπαξ ανθρωπιστική βοήθεια δεν αρκεί. Θα χρειαστεί να συνδυαστεί και με την ενίσχυση της χώρας αυτής για να αποκαταστήσει, να ανοικοδομήσει τις υποδομές της, δρόμους, γέφυρες, σχολεία κ.ο.κ. Και να ανοιχτούν περισσότεροι δρόμοι του Πακιστάν για τις εξαγωγές του Πακιστάν, για τη συμμετοχή του στο διεθνές εμπόριο κλπ. Αυτά μπορούν να αλλάξουν τον ρούν της ιστορίας και στη χώρα αυτή. Αυτά θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους οι Υπουργοί. Ευχαριστώ πολύ. Η γενικότερη αντίληψη που έχει η παγκόσμια κοινή γνώμη, αλλά και εμείς, είναι πως η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας ε, για να αντιμετωπίσει αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή στο Πακιστάν ήταν αργή και αδύναμη. Φτάσαμε καθυστερημένα και χωρίς αρκετό υλικό ή τουλάχιστον όχι με τόσο εξοπλισμό και υλικό όσο είχαμε προσφέρει σε άλλες ανθρωπιστικές καταστροφές. Και δεν καταφέραμε να καλύψουμε τις ανάγκες τις οποίες διαπίστωσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Κάποιοι Κάποιοι συνάδελφοι είπαν πως ίσως δεν υπάρχει συμπάθεια στις χώρες μας λόγω καθεστώτος στο Πακιστάν ή λόγω άλλων προβλημάτων της χώρας. Εμείς όμως ως ευρωβουλευτές θα πρέπει να προσπαθήσουμε στις δικές μας κοινωνίες να εξηγήσουμε πώς βοηθάμε ανθρώπους άτομα και όχι πολιτικά καθεστώτα. Πως η ανθρωπιστική βοήθεια βασίζεται στην ουδετερότητα, στην αμεροληψία, στην ανεξαρτησία και πως αυτές είναι οι αξίες οι οποίες εμπνέουν τη δράση μας. Στη διαδικασία Catch the Οι συνάδελφοι θα πάρουν το λόγο ε, να ξέρουν ότι είναι για ένα λεπτό η παρέμβασή τους. Η κυρία Μπασέσκου παρακαλώ. Για τον απολογισμό των ε, πλημμύρων στο Πακιστάν οφείλω να ομολογήσω ότι είναι φοβερός 2.000 άτομα έχασαν τη ζωή τους, πάνω από 2 εκατομμύρια σπίτια έχουν καταστροφεί, πάνω από 12 εκατομμύρια ζητάνε τη βοήθειά μας, ε, οι υποδομές ε, έχουν καταστραφεί, ε, πρέπει να, δεν υπάρχει τίποτα στη θέση του και Πρέπει να σας πω ότι και χώρες πιο κοντά από το Πακιστάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισαν αντίστοιχα προβλήματα αυτό το καλοκαίρι. Παραδείγματο χάρη η Ρουμανία και εμεί είχαμε πλημμύρε και μας δόθη βοήθεια 230 εκατομμύρια ευρώ. Ε, μάλλον 230 έχουν δοθεί στο Πακιστάν και είμαστε ο βασικό δωρητή. Ε, βέβαια η κατάσταση είναι καταστροφική και οι συνέπειε είναι μακροπρόθεσμε. Επομένως, ε, πιστεύω ότι μονάχα με την ε, οικονομική ανάπτυξη του Πακιστάν του ιδίου ε, μπορεί να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τραγωδία του Πακιστάν ήταν άμεση μεν, αλλά όχι ιδιαίτερα ορατή Δείξαμε την ε, αλληλεγγύη μας με τα θύματα βέβαια, αλλά 18 εκατομμύρια άτομα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν κινδύνους ε, ασθενειών και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν εισπράξει αυτή τη στιγμή μόνο το 1 τρίτο των ε, χρημάτων που είναι απαραίτητα. Και αυτό γιατί, γιατί υπάρχουν κάποιες καχυποψίες απέναντι στην διαφθορά, την, της διοίκησης στο Πακιστάν. Θα πρέπει δηλαδή να φροντίσουμε η βοήθεια αυτή να διοικητευτεί στα άτομα τα οποία έχουν ανάγκη και όχι να παραμείνουν στα χέρια των κυβερνώντων. Επίσης η ασφάλεια του, των εθελοντών που πάνε εκεί ε, πρέπει να είναι μια προτεραιότητα για μας. Για ένα λεπτό. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Κυρίες και κύριοι, καθιστάμεθα μάρτυρες μιας άνευ προηγουμένου καταστροφής στο Πακιστάν και οι άνθρωποι αν έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας. Αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι υπάρχουν περιοχές στο Πακιστάν όπου η κεντρική κυβέρνηση δεν προσφέρει καμία βοήθεια. Όπως η Πάκισταν, βόρεια του Κασμίρ και μέσα στην επικράτεια του Πακιστάν που έχει πληγεί βαριά από τις συνέπειες των πλημμυρών. Το Κίρκι Πάντισταν είδε να χάνονται 500 ζωές και ε, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων αστέγους. Έχουν απομονωθεί ολόκληρες περιοχές. Μέχρι τώρα η βοήθεια που έχει φτάσει σε αυτή την περιοχή ανέρχεται σε 10.000 ευρώ. Αυτό είναι σημαντικό τα χρήματα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να τα εμβάζει μονάχα στην κεντρική πακιστανική κυβέρνηση. Θα πρέπει τα χρήματα αυτά να, γίνει, να υπάρξει φροντίδα ώστε να φτάσουν μέχρι εκεί που χρειάζονται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, που μου δίνετε το λόγο. είναι τεραστίων διαστάσεων η κρίση στο Πακιστάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε και έδρασε πλέον αποτελεσματικά από ό,τι στο παρελθόν και αυτό μας ικανοποιεί όλους. Βλέπουμε δηλαδή ότι γίνεται πρόοδος, κυρίως σε σύγκριση με την βοήθεια που χορηγήθηκε στην ΑΕΤ. Εδώ επιθυμώ να τονίσω δύο πράγματα. Πρώτο, την ανάγκη βελτιώσεως της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν τίθεται θέμα χορήγησης ανθρωπιστικής βοήθειας. Το μέγα θέμα εδώ είναι η ανάγκη βαριών μεταγωγικών αεροσκαφών. Είναι απαραίτητα αυτά για να μεταφερθούν, να μεταφερθεί το υλικό της βοήθειας και χρειάζεται βεβαίω καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων που ε, βρίσκονται επί τόπου. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ ειλικρινά για όλα αυτά τα ε, χρήσιμα σχόλιά σας. Θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις απαντήσεις μου για τρία βασικά θέματα. Το ένα αφορά τις προτεραιότητες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες και πόσο μπορούμε να εντάξουμε την, τα σχόλια τα οποία κάνατε. Δεύτερο, πολιτικό περιβάλλον και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ουδετερότητα ε, των κοινοτικών εργαζομένων ε, και τρίτον ποια είναι η ικανότητα ε, απάντησης της κοινότητας σε θέματα επίγοντα. Το ε, για το πρώτο θέμα πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλια τα οποία ακούστηκαν σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτούς που κινδυνεύουν να αποκλειστούν και στις πιο συντηρητικές περιοχές του Πακιστάν τα άτομα αυτά είναι οι γυναίκες, και τα παιδιά, τα παιδιά που ζουν μαζί με γυναίκες, είναι, σε, είναι ομάδες υψηλού κινδύνου, οι μειονότητες, ακούστηκαν και τα θέματα των θρησκευτικών μειονοτήτων. Αυτό σε κάθε χώρα και στη συγκεκριμένη περίπτωση και στο Πακιστάν είναι ένας κίνδυνος. Οι κοινότητες αυτές που, είναι δύσκολες, που έχουν δύσκολη πρόσβαση και που είτε η φύση τους έχει αποκόψει είτε είναι απομονωμένοι λόγω συγκρούσεων. Πρέπει να σας πω ότι εξετάζουμε πάρα πολύ προσεκτικά τις προτάσεις που μας υποβάλλουν οι εταίροι μας, έτσι ώστε αυτό το οποίο χρηματοδοτούμε σε ένα μεγάλο βαθμό να στοχεύει ε, τις ανάγκες αυτών των ατόμων που κινδυνεύουν να αποκλειστούν. Και θα απαντήσω πιο συγκεκριμένα για το προσωπικό μας ε, όταν απαντήσω στη συγκεκριμένο ερώτημα για τις θρησκευτικέ μειονότητες. Ε, εξετάσουμε το θέμα των μειονοτήτων πάρα πολύ προσεκτικά και είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προφορίες για το θέμα αυτό, αλλά και για το θέμα του Κασμίρ. Και εδώ εργαζόμαστε με διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων. Επίσης, ακούστηκε το γεγονός ότι η γεωργία αποτελεί την πηγή εισοδήματος, κυρίου εισοδήματος ενός μεγάλου αριθμού κατοίκων του Πακιστάνα. Και το πρόβλημα είναι ότι πρέπει για να βελτιώσουμε την, για να βελτιωθεί κατάσταση να είμαστε επιτόπου εκεί για να βοηθήσουμε τους γεωργούς και μακροπρόθεσμα εάν, εάν διορθωθεί η κατάσταση της γεωργίας θα βελτιωθεί και το θέμα της ασφάλειας. Μακροπρόθεσμα όλα αυτά βέβαια. Τώρα, το να μπορούμε να συγκεντρώσουμε πόρους και από άλλους, δηλαδή εμείς να αποτελέσουμε την φωνή που θα ξυπνήσει τη συνείδηση των γειτόνων για να συγκεντρωθούν περισσότερα χρήματα για το Πακιστάν. Πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε άμεσα και έχουμε τώρα την ικανότητα να ζητήσουμε και τη βοήθεια άλλων. Και θα το κάνουμε αυτό τώρα που προετοιμάζουμε τη συνάντηση των φίλων του Δημοκρατικού Πακιστάν στις 14 και 15 Οκτωβρίου. Η η Βαρόνι Άστον με τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν και εγώ θα προεδρεύσουμε αυτή τη συνάντηση και θα έχουμε και μια διευρυμένη συνάντηση έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιστήσουμε την προσοχή των άλλων και να αναγκάσουμε αν θέλει να πείσουμε τους άλλους να συνεισφέρουν. Τώρα όσον αφορά τα κράτη-μέλη και όσον αφορά τους ιδίους τους δικούς μας σπόρους, τα δικά μας χρήματα, να σας πω ότι για τα 70-70 εκατομμύρια έχουν ήδη δεσμευθεί. Και ένα μεγάλο ποσό από, αυτό τον, από αυτά τα 70 εκατομμύρια έχει εκταμιευθεί. Όταν, ήμασταν στο Πακιστάν, όταν ήμουν στο Πακιστάν είχαμε ξεμείνει από χρήματα όσον αφορά τα επίγοντα ήμασταν στο πακισταν ειχαμε ξεμεινει απο χρηματα οσον ε, αφορα τα οποία εφαρμόζαμε με αξιόπιστα άτομα επιτόπου. Και το προσωπικό μας εκεί έχει καταστήσει σαφές ότι χρειάζεται περισσότερο, περισσότερα χρήματα. Πρέπει να δώσουμε και άλλα χρήματα. Τώρα, όσον αφορά τα κράτη-μέλη, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Σουδία είναι οι μεγαλύτεροι δωρητές και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω. Και έχουν δώσει τη βοήθειά τους και εμείς βέβαια από την πλευρά της Κομισιόν ε, ούτως ή άλλως είναι, είναι, είναι, ε, είμαστε συναρμόδιοι αν θέλετε, είναι μοιρασμένη η αλλως ειναι ειναι ειναι ειμαστε συναρμοδιοι αν θελετε ειναι μοιρασμενη η αρμοδιοτητα με τα κράτη-μέλη. Έχουμε συν, κοινή αρμοδιότητα με τα κράτη-μέλη στον τομέα αυτό. Θέλουμε να συνεργαστούμε και θέλουμε όλες μας οι δεσμεύσεις ε, και οι υποσχέσεις να υλοποιηθούν. Τώρα, για τα μακροπρόθεσμα, τις μακροπρόθεσμες απαντήσεις, να σας πω ότι είναι σαφές ότι οι προβλέψεις για το Πακιστάν δεν καλές. Τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Δηλαδή η πρόβλεψη για την ανάπτυξη θα αναθεωρηθεί προς τα κάτω. Από 4-5% που ήταν ε, πριν, τώρα θα πάει στο 1% για να μην πω και κάτω από το 0% και υπάρχει και άλλη μια τεράστια καταστροφή η οποία θα πρέπει να αξιολογηθεί και να εκφραστεί σε αριθμητικά στοιχεία που θα είναι δισεκατομμύρια. Αλλά θα πρέπει να κινητοποιήσουμε μια ε, σφαιρική βοήθεια για το Πακιστάν. έξω και θα πρέπει να εξετάσουμε κάθε εναλλακτική πρόταση για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Η Κομισιό βέβαια δεν έχει τη δυνατότητα να ε, δανείσει χρήματα, ε, επομένως εμείς εδώ δεν έχουμε πολλά περιθώρια από πλευρά τη Κομισιόν, όμως είναι μια εναλλακτική λύση να εξετάσουμε ποιε είναι οι ικανότητε οι του Απακιστάν και η φωνή σας θα ακουστεί όταν το συζητάμε όλα αυτά τα θέματα. Επίσης ε, υπάρχει και το θέμα του εμπορίου. Η Επίτροπος Δεκούκτ εξετάζει πάρα πολύ προσεκτικά την ε, το τι μπορούμε να προσφέρουμε στο Πακιστάν για να συνεισφέρουμε, δηλαδή, αν θέλετε, σφαιρικά στην επίλυση των προβλημάτων της χώρας. Τώρα περνάω στο επόμενο σημείο. Α, και κάτι άλλο να προσθέσω. Επίσης θα πρέπει να συνεργαστούμε με το Πακιστάν για να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση στις μεταρρυθμίσεις που έχει ξεκινήσει έτσι ώστε η οικονομία να στηριχθεί σε πιο στέρες βάσεις. Θα πρέπει να δούμε πώς χρηματοδοτούν τον προϋπολογισμό τους. Δεν θα πρέπει μέσω των, πλη, ε, πλημμυρών να καταστραφεί η κυβέρνηση. Το να βοηθήσουμε τους Πακιστανούς είναι επίσης και ένα θέμα που ε, θα εξασφαλίσει και την πολιτική σταθερότητα της χώρας αυτής. Πολιτική σταθερότητα που είναι σημαντική όχι μόνο για το Πακιστάν αλλά και για όλες τις χώρες της περιοχής. Εξού και ελπίζουμε ότι η συλλογική μας προσπάθεια ουχή μόνο θα σώσει ζωές, αλλά και θα αποφύγει την, ε, τη δημιουργία χάους στην περιοχή. Και για μάσα ε, που μας ε, αφορά το θέμα της δημοκρατίας, και ε, των, ε, των, ε, και ανθρωπιστικών ενεργειών να σας πω ότι τονίζουμε ότι για μας σημαντικό στοιχείο για την βοήθεια είναι η, εξασφάλιση της ασφάλειας των όσων ασχολούνται με την ανθρωπιστική βοήθεια. Η ουδετερότητα και η ασφάλεια των εργαζομένων στο, την ανθρωπιστική βοήθεια είναι ζωτική σημασία για μα. Υπάρχει, στις 19 Αυγούστου που είναι η μέρα για, τις, ε, για τους για τους εργαζόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα ε, τονίσαμε το γεγονός ότι έχουν χαθεί ζωές. Δύο άτομα έχασαν τη ζωή στο Πακιστάν εν μεταξύ. Δεν θέλουμε να χαθούν άλλες ζωές προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε την κρίση και την καταστροφή αυτή. Άρα τα θέματα ασφάλειας για τους εργαζομένους για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επίσης να σας πω ότι ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους σας που σχολιάσατε θετικά όλα όσα έχουμε κάνει έτσι ώστε να ε, εξασφαλίσουμε καλύτερη οργάνωση και συντονισμό. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Και θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα το τι σημαίνει συντονισμός για την περίπτωση του Πακιστάν. Όπως σας είπα, στείλαμε τις ομάδες ε, συντονισμού επιτόπου. 12 κράτη-μέλη έστειλαν ανθρωπιστική βοήθεια σε είδος. Οργανώσαμε τέσσερις πτήσεις ευρωπαϊκής αερογέφυρας προς το Πακιστάν δύο η Τσεχία, μία χρηματοδοτήθηκε από τη Φιλανδία, εφτά συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και με τον τρόπο αυτό στείλαμε βοήθεια από πολλές χώρες με συντονισμένο τρόπο στη χώρα αυτή. Και βεβαίως μοιράστηκε και επιτόπου με συντονισμένο τρόπο. Άρα λοιπόν έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο. Για όσους λένε πως θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα, θα απαντούσα ήθε να εισακουστείτε. Και θέλουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είμαστε πιο δυναμικοί στην απόκριση που δίνουμε σε τέτοιου είδους ανθρωπιστικές καταστροφές. Αυτή είναι μια συζήτηση που θα γίνει στο μέλλον και μπορώ να το συνοψίσω τη συζήτηση αυτή ως εξής. Πρώτα απ' όλα, καλύτερος προγραμματισμός. Δεύτερον, προαποφασισμένα κονδύλια από τα κράτη-μέλη που θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη στιγμή που θα ξεσπάει μια καταστροφή. Γιατί αυτή τη στιγμή όταν σημειωθεί μια καταστροφή, εγώ κάνω μερικά τηλεφωνήματα, απευθύνω μια έκκληση, αλλά δεν ξέρω τι θα μου διατεθεί. Πρέπει να σου πω ότι μέχρι στιγμή, όποτε έχω απευθύνει τέτοια έκκληση, τα κράτη-μέλη προσφέρθηκαν. Αλλά θα ήταν πολύ πιο συνετό να έχουμε ήδη από πριν στη διάθεσή μας τα κονδύλια που έχουν δεσμεύσει προς αυτή την κατεύθυνση τα κράτη-μέλη. Τρίτον, ενισχυμένο συντονισμός. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Θα πρέπει να είμαστε 27 συνένας οι οποίοι θα αντιδρούν ενιαία. Και τέλος μια πολιτική προσέγγιση στις κρίσεις αυτές, πρόληψη, οικοδόμηση, αποκατάσταση, ευθύνη. Αυτά έχω να παρουσιάσω και θα υποβάλω ως προτάσεις αργότερα σε εσάς. Και σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τα αξιότιμα μέλη για τις ε, συμβουλές και τα σχόλια προς εμένα και την ομάδα μου. Η συζήτηση έλεξε εδώ. Thank you, Mrs. Commissioner. Ε, το επόμενο μας θέμα τώρα είναι η έκθεση όρη, κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών. Ε,